καθίσετε στις θέσεις σας. Ψηφίζουμε την πρώτη έκθεση. Ψήφισμα για τη Ζιμπάμπουε. Το υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Τάι Τσαμάρα, παράγραφος 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και σας ευχαριστώ. Τώρα πάμε στο επόμενο ψήφισμα για την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια και του ομαδικού Στάφου στην Ταϊλάνδη. Παραγράφος πρώτη, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Μου ζητήθηκε να επαληθεύσω. Επαληθεύουμε λοιπόν την τροπολογία 2, παράγραφο 1. Τροπολογία 2, παράγραφος 1, εψηφίζαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και σας ευχαριστώ. έπρεπε και εγώ να κάνω την απολύθευσή μου. Δείχνουν μεγάλη προσοχή οι υπηρεσίες. Πάμε λοιπόν στροπολογία 3 υπέρ διανατάσεως. Κατά. Αποχές. Αυτό πρέπει να το επαληθεύσουμε. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία πρώτη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ευχαριστώ να επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Στο ψήφισμα, στο σύνολό του, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, είναι προφανές. Και σας ευχαριστώ. Ψήφισμα για τη Βαζιλάνδη η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Παράγραφος 9 σε δύο τμήματα, ονομαστική ψηφοφορία και στα δύο. Ξεκινούμε με το πρώτο τμήμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τη λογική σκέψη και αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, άποχες. Εγκρίνεται τη λογική σκέψη L, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία περιθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Το ψήφισμα στο σύνολό του ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και σας ευχαριστώ. Έκθεση Ντανζάν, εφαρμογή της κοινή πολιτικής άμυνας και πολιτικής ε, ε, ασφάλειας και άμυνας. Πρώτο κομμάτι, στα δύο τμήματα υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος υπαριθμών 2 ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Περάρφος Παράρφος δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστικά, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. μόνο 1. Τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η... Το αρχικό κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπέρθυμων 3 ονομαστικά. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 4 ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη τροπολογία 5 ονομαστικά. Αρχίζουμε. Πέρασε. Απερίφθη. Έχετε κάποιο πρόβλημα, πολύ φασαρία εδώ στην αίθουσα, αγαπητοί συνάδελφοι. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Με ακούτε. Πρόεδρε, δεν ξέρω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι και αν και εκείνοι παραπονιούνται, αλλά βλέπω να μην ψηφίσαμε την τροπολογία υπαριθμών 8, εκτός και αν απεσήρθη. Τροπολογία λέει ο μιλητής, μάλλον ή παράγραφο. Αγαπητοί συνάδελφοι, το αρχικό κείμενο της τροπολογίας, α, της παραγράφου 8, καταπίπτει επειδή εγκρίθηκε η τροπολογία 1 του ΕΛΚ. Είναι σαφές αυτό. Ωραία. Έχει και άλλος άνθρωπος ερώτηση. Ναι, εντάξει. Διευκρινίστε και μεν η σύγχυση, αλλά δεν μας είπατε εκείνη την ώρα ότι κατέπιπτε και γι' αυτό ψηφίσαμε προς άλλη κατεύθυνση για την τροπολογία 3 από ό,τι θα είχαμε ψηφίσει κανονικά. Μέα κούλπα αγαπητοί συνάδελφοι, εάν συμβαίνει αυτό. Αλλά είναι σαφές ότι αν εγκριθεί μία τροπολογία, καταπίπτει το αρχικό κείμενο. Για το μέλλον θα το έχω πάντα υπόψη μου και θα το επαναλαμβάνω όταν υπάρχει θέμα να καταπέσει η τροπολογία. Και τώρα πάω στην τροπολογία 6 ονομαστικά, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Παράγραφος 23 του αρχικού κειμένου. Καταπίπτει. Όχι, τα ξαναλέω γιατί μπερδεύτηκα εγώ. Προχωρώ τώρα στην ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Όχι, με συγχωρείτε. Θέλετε το λόγο. Θα ξεκινήσουμε από την 9 γιατί μπερδευτήκαμε. Αρχίσαμε με την 9, ήρθε αποσυρθεί 8. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Just to be very clear. Για να είμαστε σαφείς, το ζήτημα της παραγράφου 8 διευκρινίστηκε, αποσαφινίστηκε. Όλες οι άλλες ψηφοφορίες ήταν ονομαστικές. Τώρα είμαστε στην παράγραφο 23 η τροπολογία υπαριθμών 6 έχει καταπέσει, άρα ψηφίζουμε επί του αρχικού κειμένου της παραγράφου 23, διανατάσεως, υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 24, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 25 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. Παράγραφος 34, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της 38 ονομπέρ. Πέρασε. εγκρίνεται υπαριθμών 7 τροπολογία ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Ονομαστικά. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 43 αρχής ψηφοφορία. Ονομαστικά. Πέρας. Εγκρίνεται παράγραφο 47 αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται παράγραφο 48 σε δύο τμήματα. Υπέρ, ε, το πρώτο τμήμα, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 50, ονομαστική ψηφοφορία, αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Παράγραφος 51. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 52. Ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας, Εγκρίνεται 54, παράγραφος 54 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και ευχαριστώ συνάδελφοι. Και τώρα έχουμε την έκθεση και ευχαριστούμε τον εισηγητή. Έχουμε την έκθεση Κουκάν και Ταράντ. Χρηματοδότηση κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Πάροφο πρώτη σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην παράγραφο, παρακαλώ, ναι, θέλετε να ελέγξουμε το τέταρτο τμήμα Τη παραγράφου 1, ωραία, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3, 5 τμήματα, πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το τέταρτο τμήμα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 17. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 18. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Συγγνώμη. Τι θέλετε. Θέλετε το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Όχι. Είναι σαφές νομίζω. Συνεχίζουμε λοιπόν. Παράγραφος 19, δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται παράγραφος 28 ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά τώρα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ και περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Γκόμες για τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη, παράγραφος 1 σε δύο τμήμα πρώτο. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστικά, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14, ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Β. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, αγαπητοί συνάδελφοι, και περνάμε στην έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία. Κυρία Πύρη, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω αναβολή της ψηφοφορία για την Ολομέλεια του Ιωνίου, διότι είχαμε μία εβδομάδα μεταξύ της ψηφοφορία στην Επιτροπή και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια και πολλές νέες τροπολογίες, οπότε νομίζω είναι προς το συμφέρον και όφελος όλων των πολιτικών ομάδων, καθότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση για την Τουρκία συγκεκριμένα. Να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να ψηφίσουμε σωστά. Θα πρότεινα λοιπόν αναβολή της ψηφοφορία για τον Ιούνιο. Thank you. Ευχαριστώ. we εκφραστή υπέρ. Υπέρ, επαναλαμβάνω. Θα θέλω να μιλήσει υπέρ αυτής της πρότασης. Κυρία Πρόεδρε, είναι λογική η πρόταση νομίζω. Εντατικά και επί πέντε μήνες εργαστήκαμε πάνω στην έκθεση αυτή, αλλά η απόσταση, η χρονική ε, απόσταση ανάμεσα στην ψηφοφορία, στην Επιτροπή και την Ολομέλεια είναι τόσο σύντομη που δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε στις συμβαστικές εκείνες λύσεις που θα ήταν τόσο απαραίτητε. Γι' αυτό παρακαλώ να υποστηριχθεί το αίτημα της κυρίας εισηγήτριας. Ευχαριστώ κύριε Λάμστορφ. Ε, υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει κατά της προτάσεως. Μάλιστα. Έναν μόνο μπορώ να δεχθώ κατά Ναι, εγώ περίμενα να μιλούσε και κάποιος από τις μεγάλες ομάδες κατά της πρώτας αναβολής. Είναι πολύ σημαντικό θέμα η Τουρκία. Έχουμε ευθύνε εναντί των ψηφοφόρων μας, οι οποίοι ε, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι θέσεις έχουμε εναντί της Τουρκίας. Και πρέπει να γίνει η ψηφοφορία τώρα, να μην προσπαθήσουν να ξεφύγουν ορισμένοι. Καλώς λέει Πρόεδρος, ψηφίζουμε τώρα για την αναβολή. Υπέρ της αναβολής. Κατά αποχές και εγκρίνεται. Αναβάλλεται λοιπόν η ψηφοφορία για την έκθεση προόδου της Τουρκίας. Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώνονται έτσι οι ψηφοφορίες. Και περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου εφόσον αποχωρήσουν ε, συνάδελφοι που δεν θέλουν να παραμείνουν.